Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε με τη διημερίδα μας. Κατά την πρώτη ώρα θα σας μιλήσω ουγγρικά. Την πρώτη μου μητρική και μετά σλοβακικά τη δεύτερη. Θέμα υπαριθμών ένα στην ημερήσια διάταξη, έγκριση της ημερήσιας. Ο κύριος Μαριάς δεν θα παρίσταται σήμερα, γι' αυτό θα μεταφερθεί στις 9 Νοεμβρίου το θέμα μόνο 10. Κανένας δεν έχει αντιρρήσεις. Υπάρχουν άλλα ερωτήματα σε σχέση με το προσχέδιο. Εάν όχι, εγκρίνεται. Στη συνέχεια έχουμε την έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων. Είχαμε δύο συνεδριάσεις στις 13 και 14 Ιουλίου και τα πρακτικά της 8ης Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν αντιρρήσεις στα πρακτικά παρακαλώ των συνεδριάσεων αυτών. Διαφορετικά θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Θέμα υπαριθμών 3. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε νέους συναδέλφους, καταρχήν τον κύριο Πιέρο Σουάβε, ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά του, καθώς και τον Αλεσάνδρο Ντάβολη, που είναι δύο νέοι διοικητικοί υπάλληλοι και την Κάτια Βάτερ. Από τη Γραμματεία θα ήθελα να καλωσορίσω τα, τους υπαλλήλους αυτούς σας καλωσορίζουμε και προσμένουμε σε μια πολύ καλή συνεργασία. Στα διάφορα, εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω. Δεν υπάρχουν σχόλια και από τους συναδέλφους. Άρα εντάξει, τελειώσαμε και με τα διάφορα. Στη συνέχεια έχουμε μια αναφορά από την Ιταλία υπαριθμών 1962-2014. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν από όσο γνωρίζω. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην Επίτροπη. Κάρπεντερ ή Χαμερ, δεν ξέρω ποιος από τους δύο. Ευχαριστώ και καλό σας απόγευμα συνάδελφοι. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε το θέμα εμβριθός σε σχέση με τον κύριο Μπεράρντι, ο οποίος ε, το στην Ισημερινή Γουινέα μέχρι το Μάιο του 2015. Αυτό το θέμα σχετίζεται και με την προσωπική του μαρτυρία, αλλά και από το Human Rights Watch και διάφορες οργανώσεις των ΗΠΑ σε σχέση με ανησυχητικά στοιχεία. Εξ ονόματος της ΕΙΕΔ και εκπροσωπώ και τη Γενική Διεύθυνση ε, Justice, η οποία θα συμπληρώσει τα σχόλιά μου, θα ήθελα όμως να βασιστώ σε δύο πτυχές του ζητήματος. Καταρχήν τον χειρισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση του, της υπόθεσης, καθώς και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην η σημερινή Γουινέα. Σε δύο επιστολές που απεστάλησαν προς την οικογένεια του κυρίου Μπεράρντι, τον Απρίλιο του 2015 και μία άλλη σε οργανώσεις κοινωνίας ε, των πολιτών της Ένωσης Χριστιανών για την κατάργηση των βασανιστήριων. Σκεγραφίσαμε την προσέγγιση μας και ίσως τα γνωρίζετε ότι τα θεσμικά όργανα δεν έχουν αρμοδιότητες για την προστασία μεμονωμένων πολιτών. Πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα και υπάρχουν και οι ειδικέ διευθετήσεις για τις οποίες θα, μιλήσει, θα μιλήσουν οι συνάδελφοι τη στιγμή που δεν μπορούν οι προξενικές ή διπλωματικές αρχές να αντιμετωπίσουν, να χειριστούν το ζήτημα, διότι η Ιταλία δεν έχει γραφεία στην η σημερινή Γουινέα, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στη Λιμπρεβίλ, στην Καμπόν, καθώς και στο Καμερούν έχουμε γραφεία. Πέρα από το θέμα των προξενικών ευθυνών, είχαμε επαφές άτυπες και μη με τις επίσημες αρχές της σημερινής Γουινέας. Ε, ήρθαμε σε επαφή και στις Βρυξέλλες και στο Μαλάμπου μέσω Λίμπρεβιλ και κατά τις συζητήσεις εκείνες επιμείναμε ως προς την τήρηση των διεθνών κανόνων σε σχέση με την κράτηση καθώς και την εγγύηση των δικαιωμάτων του κυρίου Μπεράρντι για να, λάβει, να έχει ιατρική παρακολούθηση όπως πρέπει. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κράτησης είναι ένα ζήτημα που μας ανησυχεί γενικότερα. Η υπόθεση του κυρίου Μπεράρντι δεν είναι και η μόνη που μας απασχολεί σε σχέση με θέματα δικαιοσύνης, καθώς και μεταχείρισης κρατουμένων και συνθήκων κράτησης. Υπήρξε και πολιτικός διάλογος με τις αρχές της σημερινής Γουινέας και θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση εκεί είναι κάπως ασυνήθιστη. Η χώρα αυτή δεν έχει κυρώσει τις αναθεωρημένες συμφωνίες Κοτονού και δεν έχουμε τις ίδιες πολιτικές σχέσεις με τη χώρα αυτή όπως ισχύει με άλλες χώρες ΑΚΕ και με γειτονικές χώρες στην Κεντρική Αφρική. Δεν έχουμε αντιπροσωπεία εκεί και δεν χρηματοδοτούμε άμεσα την σημερινή Γουινέα. Η μη κύρωση Τη Συμφωνίας του Κοτονού σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολιτικά μέσα που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και θα ήθελα να τονίσω την πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει νομική βάση όπως θα ίσχυε σε άλλες ε, ε, περιοχές και χώρες όπως το Σαντομέ, την Γκαμπόν και το Καμερούν. Ενθαρρύνουμε την χώρα αυτή να μην απομονωθεί και προτρέπουμε τη χώρα να κυρώσει τη συνθήκη του Κοτονού έτσι ώστε να υπάρχει η βάση αντιμετώπισης ζητημάτων πολιτικής υφής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχαμε και τις ε, προεδρικές εκλογές και δυστυχώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τον εκδημοκρατισμό της χώρας, θεωρούμε ότι θα επέλθουν βελτιώσεις έτσι ώστε η σημερινή Γουινέα να μπορέσει να βελτιώσει την εικόνα της στο διεθνές προσκήνιο και να έχουμε και έναν καλός διαρθρωμένο διάλογο με τη χώρα χρησιμοποιώντας και την κοινωνία των πολιτών για υποστήριξη. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο από την Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριε Κάρπεντερ. Ο συνάδελφός μου ήδη σας και αγράφησα τα βασικά. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα για να παρέχει η ίδια προστασία. Η ευθύνη είναι στα κράτη-μέλη. Αυτά πρέπει να εξασφαλίσουν την προστασία των πολιτών τους στη συνθήκη. Έχουμε το άρθρο 23, μιλώ για την ε, συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το άρθρο προβλέπεται αρμοδιότητα, ενδεχομένως και λέγεται σε αυτό το άρθρο ότι κάθε πολίτης της Ένωσης, την επικράτη μιας τρίτης χώρας, που δεν εκπροσωπείται το κράτο ε, μέλο το οποίο είναι υπήκο δικαιούται προστασία από τι διπλωματικέ προξενικέ αρχέ ή οδήποτε κράτο μέλου. Ε, ακριβώ υπό τι ίδιε συνθήκε όπω ένα υπήκο του ελληνικού κράτου μέλου. Με άλλα λόγια, τα κράτη-μέλη παρέχουν προξενική προστασία στι υπηκό άλλων κρατών και με τι ίδιε ακριβώ ε, συνθήκε, υπό του ίδιου όρου. Ενημερωθήκαμε λοιπόν ότι αναφέρον έλαβε προξενική συνδρομή εφόσον δεν εκπροσωπεί το σε μια τρίτη ο ίδιος από την προξενική έρχη μιας άλλης χώρας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ σωστά μας εξολογήσατε την κατάσταση. Να Παρακαλώ τώρα τους συναδέλφους. Επιθυμεί κάποιος συνάδελφος το λόγο για το θέμα αυτό. Ο... Από ό,τι φαίνεται όχι. Α, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε αλλά έφτασα καθυστερημένος και δεν άκουσα την εισαγωγή για την υπόθεση Μπερνάντι. Ε, πρέπει να πω ότι Καταλαβαίνω, ακούγοντας ε, την Κομισιόν, ότι δεν πρόκειται για ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, όμως παρόλα αυτά θεωρώ ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν ε, δεν μπορεί να ασκήσει πίεση στην σημερινή Γουινέα, τουλάχιστον να ενημερώσει τις Ιταλικές αρχές, ε, να τις προειδοποιήσει για να δουν πώς θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τον εν λόγω υπηκό τους και πώς πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, τουλάχιστον να ειδοποιηθούν οι Ιταλικές αρχές από την Κομισιόν για να εξετάσουν εκ του σύνεγγης την υπόθεση αυτή που αφορά έναν δικό του υπήκο. Υπήκο της δικής τους χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος, υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Αν όχι, θα προτείνω την εξής λύση. Η αναφορά αυτή ουσιαστικά πρέπει να κλείσει κατά την απόψή μου. Δεν έχει λόγο ύπαρξης. Βέβαια, ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να γράψουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προτείνει και ο Σμαρτά. Στην επιστολή αυτή, λοιπόν, θα μπορούσαμε να ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας απαντήσει στο πώς ε, ε, σκοπεύει να βοηθήσει για τη βελτίωση των ανθρωπίνων θεμελιωδών δικαιωμάτων στην σημερινή γουίνια. Κλείνουμε λοιπόν την αναφορά και συντάσσουμε αυτή την επιστολή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία, συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Περνάμε τώρα στην επόμενη ε, αναφορά, την υπαριθμόν 944 του 2004. Σίλα Έλλης είναι η αναφέρουσα, Βρετανικής Ιθαγένειας. Η κυρία Έλλης δεν μπορεί να είναι παρούσα για λόγους υγείας. Επομένως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να δώσουμε το λόγο που εσείς Σπάιτ, πού είστε, δεν σας βλέπω. Α, εκεί είστε, μάλιστα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Yes, thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκλεισε το πλωτικό πρόγραμμα το 2000. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ε, κάποια πληροφορία ε, για το θέμα αυτό. Είδαμε όμως προσεκτικά και μελετήσαμε τις τελευταίες πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή σας και από ό,τι φαίνεται οι συνθήκες που οδήγησαν την Επιτροπή να κλείσει το πιλωτικό εξακολουθούν να ισχύουν. Και σήμερα τι θα πει αυτό. Θα πει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε ό,τι μπορούσε, έλαβε τις απαραίτητες δράσεις ε, για την επιβολή κυρώσεων, ε, ε, το περιβαλλοντικό αυτό συμβάν είναι υπό παρακολούθηση και λαμβάνονται και τα μέτρα τα ενδεδειγμένα για το μετριασμό της μόλυνσης ε, του νερού. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες εχμές ακόμη ε, στην, ε, στα επίπεδα της μόλυνσης. Καλό είναι να εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε το εν λόγω εργοτάξιο και φαντάζομαι ότι αφού θα κλείσει πολύ γρήγορα δεν θα έχουμε και λόγο ίσως να παρακολουθούμε πλέον αυτό το τοξικό χώρο ταφής αποβλήτων. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τώρα τους συναδέλφους μου που είναι στην αίθουσα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Κύριε Κρήτον Ντάρλινγκ, από καιρό ε, ασχολούμαστε με αυτή την αναφορά από τη Βανατολική Αγγλία, τη δική μου ε, περιφέρεια. Είπε και η Κομισιό ότι λόγω ε, και το έργο των αναφερών το 2013 ε, κινήθηκε η Κομισιόν κατά ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και του φορέα εκμετάλλευση αυτού του τοξικού χορταφής αποβλήτων, το Φότμουλε Spring. Και πράγματι επιβεβαιώθηκε ότι υπήρχε αυτή η ιδέα τοξικού υγρού. Έχει συνεχίσει αυτή η κατάσταση και μολύνεται και η γύρω περιοχή και ο τροφός ορίζοντας και το, το υπέδαφος. Έχουν γίνει προσπάθειες καθαρισμού, ωστόσο ακόμη δεν είναι σαφές πόσο καιρό θα στοιχίσει να μολύνει αυτός ο τοξικός χώρος. Και ποια είναι ακριβώς και η αιτία για αυτή τη ρήπαση, για αυτές τις διαρροές. Έγινε πολλή δουλειά στην περιοχή, κάναμε πολλές μελέτες και έρευνες, εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία ως προς ε, το αίτιο ε, ή αν πρόκειτο για άπαξ φαινόμενο ήταν αποτέλεσμα κάποιας ε, παράβασης, είναι μακροχρόνιο το πρόβλημα. Δεν έχουμε καταλήξει. Η αν πρόκειται για απαξ φαινομενο ηταν αποτελεσμα Έλλης δυστυχώς ε, που θα μπορούσε να μας κάνει εδώ μια επικαιροποίηση της κατάστασης ε, δεν μπορούσε να είναι εδώ λόγω υγείας, ούτε οι άλλοι αναφέροντες λόγω υγείας και άλλων περιορισμών. Είχαμε μια συνάντηση τον Ιανουάριο μεταξύ της ΔΕΦΡΑ, του Περιβαλλοντικού Οργανισμού και των αναφερόντων, επί τόπου και καταφέραμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε, να βρούμε περισσότερες πληροφορίες για την ε, ρήπανση στο Hotness Spring. Ο φορέας θα πρέπει να εξορίξει νέα φρεάτια ε, για να δει αν πράγματι πρόκειτο ε, για ένα φαινόμενο, μόνο μία φορά δηλαδή η μόλυνση προκλήθηκε από το, πριν από πολλά χρόνια ή αν είναι κάτι που επαναλαμβάνεται ως φαινόμενο. Υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση και την ποιότητα του, της ποιότητας υδάτων από ένα παρακείμενο διοστάσιο, παίρνουμε στοιχεία. Η περιβαλλοντική οργάνωση, ο περιβαλλοντικός οργανισμός τον Ιούνιο φέτος δείχνει ότι υπάρχει πράγματι δράση, αναλαμβάνεται δράση για την ε, βελτίωση της κατάστασης ε, και κατά την άποψή μου ήδη από την αρχή ε, αυτό που θέλαμε ήταν διάθεση πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους γιατί ένα από τα βασικά προβλήματα που είχαμε με την αναφορά ήταν η έλλειψη επικοινωνίας και πληροφόρησης των αναφερόντων οι οποίοι δεν τηρούνταν ενήμεροι και αυτό δημιούργησε έλλειψη εμπιστοσύνης όπως καταλαβαίνετε και δεν υπήρχε συνεργασία μεταξύ των πλευρών. Και αυτό δημιούργησε εντάσεις και σε τοπικό επίπεδο, όπως καταλαβαίνετε. Πρόσφατα, ε, οι αναφέροντες έγραψαν ε, στην Επιτροπή μας και συγκεκριμένη κυρία Έλλης αναφέροντας την αποψή της, είπε ότι τα επίπεδα ρήπανση εξακολουθούν να είναι πάνω από τα αποδεκτά επίπεδα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και εμείς έτσι θεωρούμε ότι είναι τα πράγματα στην περιοχή αληθεύει ότι οι μετρήσεις από τα φρεάτια δείχνουν ε, ότι υπάρχει αυτό το αμμονίουχο άζωτο σε πάρα πολύ μεγάλη περιεκτικότητα ακόμη. Ε, το 2008-2010 είχαμε κάποια ατυχήματα, αλλά για μας δεν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για να ληφθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αναφέρεται και το οποίο έχουν επισημάνει. Με βάση λοιπόν όλα αυτά ε, και το ότι υπάρχει ένα τοπικό σχέδιο, αυτό που θέλουμε να προτείνουμε στην Επιτροπή Αναφορών είναι οι αγγλικές αρχές να κληθούν να μας αναφέρουν για την τρέχουσα κατάσταση αυτού του χώρου ταφής αποβλήτων και να μας πούν συγκεκριμένα τι γίνεται με αυτά τα νέα φράτα τα οποία άνοιξαν και ποια είναι οι μετρήσεις και από το παρακείμενο αντιλοστάσιο ώστε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση για να ε, επιβεβαιωθούμε ότι θα επιβεβαιώσουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα στο, των Λεσπρίνγκ. Ευχαριστώ. Στρέφομαι στους συναδέλφους. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Όχι, δεν βλέπω κανένα να θέλει να πάρει το λόγο. Οπότε πραγματικά τώρα βρίσκομαι στην ε, δύσκολη θέση να πρέπει να πάρω μια απόφαση. Η αναφορά αυτή υπευλήθη το 2004, πριν από 12 χρόνια. Και θα πρέπει όντως να δούμε το φάκελο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε 12 ε, φορές για την ε, ε, αναφορά αυτή. Είναι η 8η φορά που μπαίνει στην ημερήσια διάταξή μα η αναφορά αυτή και κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό σε βάθος. Ούτε ότι δεν του έχουμε δώσει την δέουσα προσοχή. Η πρόταση τώρα της γραμματείας μου φαίνεται λογική, αν μπορείτε να το δεχτείτε κι εσείς, να ε, παγώσουμε την αναφορά αυτή, γιατί δεν βλέπω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Βεβαίως, αν αυτό το πρόβλημα εξεκολουθήσει να υπάρχει, βεβαίως ε, μπορεί να υποβληθεί καινούρια αναφορά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ασχοληθούμε περαιτέρω με την ε, αναφορά αυτή. Μπορούμε νομίζω να την κλείσουμε. Έχουν υπάρξει κάποιες θετικές αλλαγές. Αν τώρα μπορείτε να δεχτείτε την πρότασή μας, μπορούμε να κλείσουμε τούτη την αναφορά. Αν το πρόβλημα συνεχίσει να υφίσταται, μπορεί να υπάρξει υποβολή νέας ε, αναφοράς. Γιατί τόσα χρόνια ε, εξεκολουθεί να υφίσταται αυτή η αναφορά και δεν βλέπω γιατί πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Αυτή είναι η πρότασή μου. Δεν ξέρω, οι συνάδελφοι μπορούν να συμφωνήσουν. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι έχουμε χρόνια που ασχολούμαστε με την αναφορά αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι ε, επειδή την έχουμε πολλά χρόνια στην Επιτροπή μας την αναφορά αυτή σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να την κλείσουμε. Τα προβλήματα που έχουμε στην περιοχή εξακολουθούν να υπάρχουν και ναι υπάρχει ένα πρόγραμμα εργασίας σε τοπικό επίπεδο αλλά αυτό είναι ακριβώ και ο λόγο που καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο. Γιατί είναι ακόμη ανοιχτή η αναφορά αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε αυτή την αναφορά ε, ανοιχτή τουλάχιστον για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ίσως, για να δούμε μήπως μπορούμε όντως τελεσίδικα να το λύσουμε μέσω σωστή κατάλληλη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό είναι και ο ρόλος της Επιτροπής Αναφορών, να βρει μη δικαστικούς τρόπους να λύσει προβλήματα που θίγουν οι πολίτες. Και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε, με, ενεργά φυσικά. Αλλά ένα τμήμα όλη αυτή τη ενεργού συμμετοχή σημαίνει ότι ε, προέκυψε μάλλον λόγω του ότι ακριβώς ήταν ανοιχτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η αναφορά αυτή. Η μόλυνση εξακολουθεί. Η διαρροή εξακολουθεί να υπάρχει και δεν ξέρω τώρα αν ήταν η ε, διαδικασία επιπαραβίαση, ε, επιπαραβάση συγγνώμη, επαρκής για να λυθούν τα προβλήματα. Γι' αυτό εγώ ζητώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή. δεν θέλω να προτείνω πράγματα που δεν μπορείτε να, συμφωνήσετε, γιατί εγώ σέβομαι την άποψή σα απολύτω, αλλά το θέμα δεν είναι ότι είναι μια αναφορά που χρονίζει στην Επιτροπή μας. Το είπα να την κλείσουμε γιατί δεν βλέπω τι άλλο θα μπορούσαμε πιθανώς να κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω ε, αν έχει κάτι να πει, ο κύριος Σπέιτ ίσως. υπάρχει κάτι, κάποιο μέσο που να μπορείτε εσείς να χρησιμοποιήσετε ή να μας πείτε κάτι που θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε, γιατί η Κομισιόν έχει ήδη κάνει πολλά και εμείς στην Επιτροπή Αναφορών έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε. Μπορείτε να μας πείτε κάτι άλλο που ίσως μπορούσε να γίνει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δίκιο έχετε ότι έχουμε εξαντλήσει το φάσμα των ε, ενδικών μέσων που υπάρχουν ε, διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά τώρα, αν υπάρξει μεγαλύτερη αύξηση στην ε, μόλυνση και αλλάξει η κατάσταση επιτόπου, τότε μπορούμε να αναθεωρήσουμε το φάκελο. Αλλά προ το παρόν δεν έχουμε κάποια άλλη δράση που να μπορούμε να πάρουμε, τουλάχιστον από τη δική μα τη μεριά. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την Ζουντίτ γιατί ε, εάν ε, θέλετε να κάνετε περισσότερα πράγματα και σε τοπικό επίπεδο όλα να έχουν αίσιο πέρας, θα μπορούσαμε να αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή και να δούμε πώς θα διευθετηθούν τα πράγματα ειρηνικά ή δυνατόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατανοώ ότι είναι μακρύ το χρονικό διάστημα για να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, αλλά δεν μπορούμε να την αφήσουμε ανοιχτή για λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εγώ θα μπορούσα να το υποστηρίξω αυτό. Άλλοι που θα ήθελαν το λόγο. Συμφωνώ και εγώ, Πρόεδρε, μαζί σας πιστεύω ότι πρέπει να κλείσει αυτή η αναφορά. Γιατί αν την αφήσουμε ανοιχτή δεν θα έχουμε κάποια αίσια έκβαση. Νομίζω ότι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση θα ήταν να γράψουμε στις αρχές της Μεγάλης Βρετανίας και να ζητήσουμε τις πληροφορίες σε σχέση με τα φρεάτια αυτά. Μετά θα δούμε κατά πόσο υπάρχει επιβεβαίωση και αν η κατάσταση είναι σταθερή και αν έχει επιληθεί τοπικά το ζήτημα από ό,τι μας είπε και η βουλευτής και στο μέλλον να κλείσουμε την αναφορά αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε πληροφορίες για τα νέα φρεάτια αυτά. Θέλουμε να δούμε πώς έδρασε η κυβέρνηση, ο ιδιωτικός τομέας και οι τοπικές αρχές. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό πριν κλείσουμε αυτή την αναφορά. Προσπαθώ να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, όπως καταλαβαίνετε. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν σήμερα. Δύο συνάδελφοι συμφωνούν μαζί σας, γι' αυτό θα μπορούσαμε να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια Εάν ανακύψουν νέα στοιχεία ή βελτιώσεις, τότε θα προτείνουμε να κλείσει η αναφορά το Δεκέμβριο. Συμφωνείτε? Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, Περνάμε στην επόμενη αναφορά, 2014 από τον Ρομπέρτο, του Ρομπέρτο Πόντσιο από την Ιταλία. Από όσο γνωρίζω, ο κύριος Πόντσιο είναι παρόν. Έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά. Εκτός μικροφώνου. Θα ήθελα να λάβετε υπόψη την αρχική αναφορά του 14 σύμφωνα με τα στοιχεία της 29ης ε, Σεπτεμβρίου του 16 γιατί εδώ βρισκόμαστε σε μία ιδιάζουσα κατάσταση. Στο μεταξύ, οι Ιταλικές αρχές παρενέβησαν. Σημασία έχει να δούμε κατά πόσο έδρασαν σωστά. Άρα στα πέντε λεπτά τηλεγραφικά θα σας πω ότι η αναφορά αυτή δεν υποβλήθηκε από έναν πολίτη. Εγώ εκπροσωπώ τέσσερις νομικές, τέσσερα νομικά πρόσωπα. Την κοινότητα της Άλμπα, την ε, ένωση της ε, καλλιέργειας της τρούφας και άλλες δύο ενώσεις και οργανισμούς. Αυτό διαφοροποιεί την Ιταλία από την, από την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί εμείς θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο το άρθρο 29 μετά από συμβιβασμό λαμβάνει υπόψη και την κοινοτική υπεροχή του δικαίου. Δηλαδή το ότι δεσπόζει το κοινοτικό δίκαιο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πρόκειται για έναν ε, νομικό συμβιβασμό που δείχνει ότι το ζήτημα δεν έχει επιληθεί. Στην Κροατία, στη Γαλλία και στην Ισπανία υπάρχει ΦΠΑ 4%. Σε εμά όμως το ποσοστό είναι 22% και μπορεί να φτάσει και το 24%. Σε σχέση λοιπόν από, σε σχέση με την ε, Ιταλική νομοθεσία δεν μπορούμε την ε, τρούφα στην υπόλοιπη Ευρώπη να τη θεωρούμε γεωργικό προϊόν, ενώ στην Ιταλία δεν αναγνωρίζεται αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι παράδοξο και παράλογο δυνάμει της νομοθεσίας μας, διότι τα μανιτάρια στην Ιταλία έχουν ΦΠΑ 4%. Η τρούφα όμως η οποία βρίσκεται στο υπέδαφος δεν θεωρείται γεωργικό προϊόν και έχει ΦΠΑ 22%. Όμως η τρούφα στην ουσία είναι γεωργικό προϊόν. Αυτό αντιτίθεται και στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πάντα θεωρούσε αυτό το προϊόν γεωργικό προϊόν. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Στην Ιταλία ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές αρχές, εκρεμεί ένας νόμος που είναι ο νόμος 1776 του 2015 και ε, δυνάμει αυτής της νομοθεσίας ο κύριος Τσόλος, επίτροπος, θεώρησε ότι η τρούφα θα πρέπει να θεωρηθεί γεωργικό προϊόν για να μην υπάρχει διάκριση δεν θα πρέπει να χάσει την ανταγωνιστικότητά του το δικό μας ε, προϊόν. Εκρεμεί αυτή η κατάσταση και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν δόθηκε συνέχεια. Έχουμε να κάνουμε με μία κατάσταση αμβλήνιας θα μπορούσα να πω σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό νόμο. Πώς είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεωρεί ότι η τρούφα είναι γεωργικό προϊόν με τους αντίστοιχους κωδικούς, ενώ δεν το δέχεται η Ιταλία. Πώς μπορεί να υπάρχει διαφορετική διαχείριση μεταξύ Γαλλίας, Ισπανίας και Κροατίας από τη μία πλευρά και ε, από την πλευρά της Ιταλίας να υπάρχει ο πενταπλάσιος ΦΠΑ. Γι' αυτό θα θέλαμε δυνάμει των άρθρων 4, ε, 39 ε, και 40 να αναθεωρηθεί αυτό το πλαίσιο. Εάν θέλετε να υπάρχει σωστός ανταγωνισμός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η αρχή. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συντονισμός. Θέλουμε σταθεροποίηση των αγορών μα φτάνουμε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Εάν θέλουμε λογικές τιμές για τον καταναλωτή θα πρέπει να λάβουμε τα αντίθετα μέτρα. Θα πρέπει να αντιστρέψουμε την κατάσταση και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δυστυχώς ε, ισχύουν ακόμα οι κανόνες που οδήγησαν στην αναφορά. Γι' αυτό θα πρέπει η Ιταλία να μην ακολουθεί μία μεμονωμένη και αμφίσιμη θέση, αλλά να ακολουθήσει την κοινοτική νομοθεσία. Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Ο κύριος Άλλη έχει το λόγο. Παρακαλώ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αρχικά η αναφορά ε, βασιζόταν στα στοιχεία της Ιταλικής ε, νομοθεσίας που αντιτίθεται στην ε, Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και γι' αυτό λάβαμε διάφορες προσφυγές. Γι' αυτό ανοίξαμε μία διαδικασία ε, διαμέσω του U-Pilot κατά της Ιταλίας για να επιλύσουμε το θέμα αυτό. Η Ιταλία αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα στην νομοθεσία της τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και η Επιτροπή θεωρεί ότι θα τροποποιηθεί η νομοθεσία, γι' αυτό η Ιταλία συμμορφώνεται με το κοινοτικό δίκαιο, δέχτηκε αυτή την τροποποίηση του νόμου και έκλεισε τη διαδικασία U-Pilot. Ο αναφέρον θεωρεί ότι το γεγονός ότι οι τρούφες υπάγονται σε ένα καθεστώς φορολογίας του 10% αντιτίθεται και αντιβαίνει το κοινοτικό δίκαιο για δύο λόγους. Γιατί υπάρχουν γεωργικά προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε ΦΠΑ 4%. Και υπάρχουν και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπάρχει φορολόγηση της τρούφας με χαμηλότερο συντελεστή. Όμως η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η απόφαση δεν αντιτίθεται στις ε, νομοθετικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί στην Ιταλία υπάρχουν πολλά είδη διατροφής και γεωργικά προϊόντα που φορολογούνται με 10%, 5% και 4%. Υπάρχουν τρεις συντελεστές. Αυτό είναι θέμα διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών που μπορούν να αποφασίσουν για τον συντελεστή ΦΠΑ τη στιγμή που τηρούνται οι αρχές της οδηγίας. Ως προς τη διαφορά συντελεστή με άλλες, σε σχέση με άλλες χώρες όπως η Ισπανία, Γαλλία και Κροατία, αυτό δεν αφορά αποκλειστικά την τρούφα. Τα περισσότερα, για τα περισσότερα προϊόντα υπάρχει διαφορά ε, συντελεστή φορολόγησης. Αυτό δεν αποτελεί πρόσκομα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και στην ανταγωνιστικότητα. Είναι θέμα φορολογικής απόφασης των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη ορίζουν του συντελεστές φορολόγησης τη στιγμή που τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, εάν πλήττεται ο ανταγωνισμός, τότε θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε. Όμως, σε αυτή την περίπτωση και με βάση την προστιθέμενη αξία του προϊόντος, μπορούμε να πούμε ότι ο συντελεστής είναι ο συντελεστής που ισχύει στην χώρα εξαγωγής. Δηλαδή, ο ΦΥΠΙΑ ορίζεται στην Ιταλία ανεξάρτητα από την προέλευση του προϊόντος, αν προέρχεται από την Κροατία, Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία. Γι' αυτό θεωρούμε ότι οι Ιταλικές αρχές επέλυσαν το ζήτημα με βάση τις αρχές που διέπουν το κοινοτικό δίκαιο. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε εσείς επιμένετε ότι αυτό είναι θέμα πολιτικο... Ε, εθνικών αρμοδιοτήτων, άρα δεν ε, έχουμε δυνατότητα ιδιαίτερης παρέμβασης ώστε να κάνουμε διαφορά. Συνάδελφοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μια γενική σκέψη για το ρόλο αυτής της Επιτροπής. Το γεγονός ότι μία αναφορά που παρουσιάστηκε εδώ οδήγησε στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου της Ιταλίας δείχνει ότι η εργασία μας είναι πολύ σημαντική, διότι μετά την υποβολή της αναφόρας από τον Ρομπέρτο Πόντσιο που εκπροσωπεί τον κόσμο της Ιταλικής ε, τρούφας η κατάσταση άλλαξε άρδιν στην Ιταλία. Όμως δεν υπάρχει πλήρης προσαρμογή. Ακούσαμε την ε, άποψη της Επιτροπής ε, που θεωρώ ότι ανήκει στην Γενική Διεύθυνση ΤΑΞ ε, που ασχολείται με το φορολογικό καθεστώς της τρούφας μεταξύ άλλων. Όμως ένα άλλο, μια άλλη πτυχή του ζητήματος αφορά τη φύση της τρούφας τον ιδιάζοντα χαρακτήρα δηλαδή της τρούφας. Δηλαδή, όταν μιλάμε για γεωργικό προϊόν σε μία χώρα και όχι σε μία άλλη, με βάση τις οργανοληπτικές ιδιότητες, η αντιμετώπιση αυτή είναι παράλογη και θα πρέπει να δούμε τι ισχύει ως προς τη φορολόγηση, ε, την πιστοποίηση του προϊόντος και ε, να λάβουμε υπόψη ότι όπου θεωρείται γεωργικό προϊόν, τότε γίνονται επενδύσεις. Όταν δεν θεωρηθεί γεωργικό προϊόν, δεν προσδίδονται αυτοί οι πόροι. Δεν αποδίδονται αυτοί οι πόροι. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη ότι η Ιταλική κυβέρνηση άρχισε αυτή τη διαδικασία προσέγγισης, και αυτό εν μέρει είναι θετικό, θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, λαμβάνοντας υπόψη και την άποψη της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη. Δηλαδή, χρειαζόμαστε και την άποψη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας. Δηλαδή, θα πρέπει να, να μας πει κατά πόσο η τρούφα την χάνει της ίδιας αντιμετώπισης στις διάφορες χώρες, Κροατία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. για να δούμε ποια είναι και τα σχετικά πλεονεκτήματα που διέπουν την, τον τομέα της ε, τρούφας σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσα στα πλαίσια ενός ε, ε, ρυθμιστικού πλαισίου. γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τρούφα έχει έναν ιδιάζοντα χαρακτήρα, ανήκει σε αυτόν που την βρίσκει και γι' αυτό θα θέλαμε την γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη. Ε, χαίρομαι που βλέπω ότι είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος ώστε να κλείσει το θέμα αυτό. Βεβαίως να ακούσουμε και άλλες απόψεις αν υπάρχουν. Δεν είμαι ειδικό σε θέματα... Δεν είμαι ειδικός σε θέματα τρούφας. Απλά αυτό που θέλω να πω έχει να κάνει πιο πολύ με τη δική μου άποψη για το τι θα έπρεπε να είμαστε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εγώ θέλω να υπάρχει μια φορολογική, κοινωνική, περιβαλλοντική εναρμόνιση και στην προκειμένη περίπτωση, όπω καταλαβαίνετε, εναρμόνιση και για τον ΦΠΑ ε, στην τρούφα. Τώρα, ε, καταλαβαίνω τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ίδια ακούμε κάθε φορά. Είναι μόνιμη αποδόση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εθνική αρμοδιότητα, όπω και ο ΦΥΠΑ, στην προκειμένη περίπτωση, Όμω όχι για τα κριτήρια οικονομική σύγκληση. Εκεί είμαστε όλοι στην ίδια σχολή, αν θέλετε, στο ίδιο σχολείο πάμε και πρέπει όλοι να είμαστε καλοί μαθητέ και να σεβόμαστε τα κριτήρια. Υπάρχει πολιτική βούληση. Τι θέλουμε ω Ευρώπη. Εάν θέλουμε ένα είδο dumping, για το κόστος της τρούφα τώρα δεν ξέρω ακριβώς ε, ποιο είναι το μερίδιο της Ιταλικής αγοράς και τα λοιπά, αλλά από εκεί και πέρα αυτά τα τόσο σπάνια και δαπανηρά μετά, τέλος πάντων υπάρχουν άλλα πράγματα που τα αφήνουμε, ίσως να υπάρχει και σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ξέρω, αλλά το να λέμε να ζητήσουμε την Επιτροπή τη Άγκρη να γνωμοδοτήσει, γιατί όχι, δεν είναι κακή ιδέα. Ε, τώρα για τους Ιταλούς παραγωγούς τρούφας, αν τελικά πάρετε 4% ΦΠΑ, θα μετακυληθεί το όφελος στον καταναλωτή γιατί στην αιστεία σημειώθηκε στη Γαλλία κατά 14 μονάδε μονάδες ο συντελεστής. Υπόσχονταν οι εστιατόρες ότι αν κατέβει ο ΦΠΑ ποτέ στο 5% θα μείωναν την τιμή των πιάτων στα εστιατόρια. Ούτε το ένα έγινε ούτε το άλλο έγινε τελικά. Ένα λεπτό κύριε Πόντζιο και θα σας δώσω το λόγο, θα σας δώσω το λόγο, ναι. Ε, απλώς να ακούσουμε και τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές σε περίπτωση που θέλουν κάτι να πούν. Όχι. Όχι. Ωραία. Ο κύριος Πόνσιο έχει το λόγο λοιπόν. Να απαντήσω ευχαρίστω στο ερώτημα. Βεβαίως, ο τελικός καταναλωτής ε, ευεργετείται. Εάν εγώ ε, είμαι εκ νέου πολιτής, δηλαδή μεταπολιτής και πρέπει να φορολογήσω κατά 10% σε σχέση με το 4% που ισχύει σε άλλες ε, χώρες, τότε φυσικά πλήττεται ο καταναλωτής. Εάν εγώ στην ε, ε, Ιταλία έχω τον ίδιο ΦΠΑ, αυτό επεργετεί τον τελικό καταναλωτή. Γι' αυτό, ακριβώς επειδή θέλουμε να προστατεύουμε τον καταναλωτή, Θέλουμε να ε, έχουμε ένα λογικό και ενιαίο ΦΠΑ και ιδιαίτερα στην περίπτωση μεταπόλησης. Το κέρδος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα φορολογείται ακόμα περισσότερο σε περίπτωση μεταπόλησης. εδώ το πρόβλημα. Δεν είναι κατά πόσο στην Ιταλία υπάρχει ένα προϊόν που θεωρείται γεωργικό ή όχι. Μιλάμε για το ίδιο προϊόν που είναι η τρούφα, το οποίο στη Γαλλία, Ισπανία και Κροατία υφίσταται μία διαφορετική μεταχείριση από ό,τι στην ε, Ιταλία. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρώπη να συντονίσει αυτή την κατάσταση, αλλιώς θα υπάρχουν συνεχείς δυσλειτουργίες. Αυτές είναι οι κοινέ αρχές ε, της Ευρώπης, δηλαδή να υπάρχουν κοινοί κανόνες και όχι αυθαίρετοι. Δεν μπορεί να αυθαίρεται μία χώρα, δηλαδή στην Ιταλία αυτό το προϊόν θεωρείται προϊόν πολυτελείας, όπως οι γούνες, ενώ στην, στην Ισπανία, Γαλλία και Προακτία θεωρείται ένα γεωργικό προϊόν. Γιατί εγώ στο Σανρέμο θα πρέπει να έχω μία διαφορετική κατάσταση από ό,τι ισχύει στο Μεντόν, δηλαδή με το που θα διαβώ τα σύνορα 20 μέτρα πιο εκεί ή αυτό αφορά την Ίστρια στην Κροατία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα μανιτάρι το οποίο βρίσκεται στο υπέδαφος. Γιατί πρέπει λοιπόν να υφίσταται φορολόγηση 4% στις άλλες χώρες και 10%, 22% στην Ιταλία. Θα πρέπει να υπάρχουν κοινοί κανόνες και κοινή αντιμετώπιση όχι διαφοροποιημένη. Δεν θα επιλύσουμε το πρόβλημα μειώνοντας ε, την ε, ζημία. Δυνάμει του άρθρου 29 ε, δεν μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα στην ολότητά του. Γιατί θα μπορούσε κανείς ε, να προχωρήσει και σε άλλες καταστάσεις που εντάξει δεν σας αφορούν εδώ. Δηλαδή αυτός που καλλιεργεί τρούφες δεν μπορεί να υφίσταται ένα διαφορετικό φορολογικό καθεστώς. Καθίσταται σαφές ότι υπάρχει, υπάρχουν διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Βεβαίως μειώθηκε η ζημία με το 10% αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν αρθεί οι διακρίσεις. Ευχαριστούμε κύριε να προσπαθήσω να συνοψίσουμε λίγο τη συζήτηση. Από τη μια, η εναρμόνιση των συντελεστών ε, ΦΠΑ είναι ένα θέμα σημαντικό. Ακούσαμε τι είπε η Κομισιόν. Και βεβαίως ε, συμφωνώ με πολλές απόψεις εγώ, αλλά είναι σημαντικό θέμα το θέμα της εναρμόνισης του ΦΠΑ και δεν ε, μπορούμε να το προσπεράσουμε. Βεβαίω, και αυτό που λέει ο κύριο Μπόντσιο είναι σημαντικό. Κατανοώ την άποψή του και εγώ καταναλώνω τρούφες. Αλλά καταλαβαίνω το ότι αυτό το προϊόν δεν θεωρείται γεωργικό προϊόν στην Ιταλία. Μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε ίσως ε, την ε, άποψη και των συναδέλφων από την Επιτροπή Γεωργίας. Θα κρατήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά αυτή και θα δούμε πότε θα την κλείσουμε, με βάση και τις επόμενες γνωμοδοτήσεις που θα λάβουμε. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο αυτό και πάμε στην αναφορά υπαριθμών 0755 του Άντζελο Αλού, Ιταλού πολίτη, σχετικά με την καθιέρωση του δικαιώματο πρόσβασης στο διαδίκτυο ως θεμελιώδους αρχής. Ο αναφέρον δεν είναι εδώ, οπότε θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τον αναφέροντα ότι η ευρυζωνικότητα, η πρόσβαση στο διαδίκτυο προσλαμβάνουν ε, όλο και μεγαλύτερη σημασία γιατί συμμετοχή στην ε, συμμετοχική ψηφιακή δημοκρατία για τη συμμετοχή στα κοινωνικά επαγγελματικά δρόμενα, αλλά και για την ε, άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης ε, και λόγου. Το 2013 λάβαμε αυτή την αναφορά. Έκτοτε έγιναν πολλά, αν δείτε και την αγορά, αν δείτε τι γίνεται στην ευρωπαϊκή αγορά ευρωζωνικότητας, υπάρχουν δυνατότητα, δυνατότητες, ουσιαστικά όλοι πια έχουν πρόσβαση σε αυτήν την τεχνολογία. Σίγουρα υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ακόμη για πολλούς λόγους δεν έχουν έχουν πρόσβαση σε ευρωζωνικά δίκτυα, αλλά και οι υψηλή ποιότητα ε, συνδέσει ε, έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί με μεγάλη προσοχή με το θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια πρόταση Μία πρόταση που λεγόταν Connected Continent, ε, πρόταση κανονισμού για τη διασύνδεση της Ευρώπης. Πέρυσι επίσης Κοινοβούλιο και Συμβούλιο συμφώνησαν με την πρόσβαση στο ανοιχτό διαδίκτυο. Άρα τα δύο τελευταία χρόνια νομίζω έχουμε καταφέρει να προωθήσουμε την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς παρακολήσεις, εμπόδια και άλλα προβλήματα για την πρόσβαση στο διαδικτυακό περιεχόμενο υπό την προπόθεση ότι υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Το Σεπτέμβριο τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ε, μια δέσμη μέτρων για την ε, συνδεσιμότητα όπως τη λέμε και εκεί περιλαμβάνονται διάφορα μέτρα και εργαλεία όπως και η αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Σε αυτό το πλαίσιο η διασύνδεσιμότητα, το connectivity στα αγγλικά, ε, είναι προϋπόθεση, όπως και οι στόχοι προώθησης ε, του ανταγωνισμού, προώθηση της εσωτερικής αγοράς κτλ. Η πρόταση οδηγίας, λοιπόν, ε, τι σκοπό έχει να βελτιώσει επενδύσεις και στο, και στη σταθερή και στην ε, ασύρματη ευρυζωνική ε, επικοινωνία, να διευκολυνθεί ακόμη δηλαδή περισσότερο η πρόσβαση στο διαδίκτυο και είναι σημαντικό να πούμε επίσης αυτό το πλαίσιο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει και εξυγχρονισμό των κανόνων για την καθολική υπηρεσία Αντί λοιπόν να ε, προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τις παραδοσιακές υπηρεσίες ε, που φυσικά βέβαια παραμένουν σημαντικές αλλά με τη νέα ε, νομοθεσία για την καθολική υπηρεσία θα ρυθμίζουμε την πρόσβαση στα βασικά ευρωζωνικά δίκτυα και θα προτείνουμε κανόνες δυνάμει των οποίων κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει συμβόλαια που θα του δίνουν πρόσβαση σε βασικά ευρυζωνικά προϊόντα, δηλαδή θα μπορεί ο κάθε πολίτης ε, μέσω της διασύνδεσης του, ε, μέσω της σύνδεσης στο διαδίκτυο να συμμετέχει πλέον, πλέον, πλήρως πλέον στην ψηφιακή κοινωνία. Έχουν γίνει πολλά λοιπόν τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε το διαδίκτυο να είναι απόλυτα προσβάσιμο και σε προσθέσεις τιμές και αυτό για όλους τους πολίτες. Εξού και καταθέσαμε, σα είπα, αυτή τη δέσμη μέτρων το Σεπτέμβριο για τη συνδεσιμότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα σημαντικό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Maybe it's a time for me to change my... Ίσως είναι ώρα να αλλάξω γλώσσα από τα ουγγρικά να περάσω στα σλοβενικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους. Ε, θέλει κάποιος να παρέμβει, να πει κάτι. Δεν είναι τυχαίο βεβαίως που άλλαξα γλώσσες ε, τώρα, γιατί η Σλοβακική Προεδρία έχει, ε, που έχει και την Προεδρία έχει δηλώσει ότι θα είναι ένα από τις, από τις προτεραιότητες της το θέμα αυτό της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει αναφερθεί και στα σημαντικά έγγραφα κλειδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι αν σε αυτή την κατάσταση έχει νόημα να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Γιατί ίσως αυτή η αναφορά να μπορούσε να κλείσει είναι στρατηγικής φύσεως το ερώτημα. Είναι θετική η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές αναφορές ε, στα διάφορα ε, έγγραφα ε, της Επιτροπής σχετικά. Οπότε, ή ε, να κλείσουμε το, ε, την αναφορά αυτή, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να το μελετά. Ο κύριος Τσίριο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Το θέμα του ευρυζωνικού και της πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι πολύ σημαντικό. Και ο συνάδελφος ε, Πολιέζε και εγώ παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την αναφορά, γιατί είναι κάτι το νέο, κάτι το καινούριο. Πρόκειται για δικαιώματα που κάποτε δεν υφίσταντο και δεν τις ε, βλέπουμε αυτές τις ε, προτεραιότητες παραδιαφορετικά σήμερα. Σήμερα μιλάμε για το ε, ευρυζωνικό. Σκεφτείτε όμως ε, τι γίνεται στις ορεινές περιοχές, εκεί που δεν υπάρχει ευρυζωνικό δίκτυο, δεν θα, αντικα, δεν θα εγκατασταθούν, με επιχειρήσεις. Θα υπάρχει λοιπόν το λεγόμενο digital divide, αυτός ο ψηφιακός διχασμός και διαφοροποίηση, κάτι το οποίο απασχολεί και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Αυτό που θέλουμε να ξέρουμε είναι κατά πόσο μέσα στα πλαίσια των νέων δικαιωμάτων αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο θα μπορούσαμε να υπερασπιστούμε και αυτό ισχύει αν λάβουμε υπόψη την ψηφιακή πραγματικότητα. Κάποιος άλλος συνάδελφος που θα ήθελε το λόγο. Ak να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και όταν λάβουμε μία απάντηση από την ΑΦΚΟ να την κλείσουμε. Σας ευχαριστώ. Εάν συμφωνείτε όλοι, λοιπόν, με αυτή την εξέλιξη θα μπορούσαμε να πούμε ότι παραμένει ανοιχτή και επιτελείται πρόοδος. Θα προσεγγίσουμε τους συναδέλφους από την Επιτροπή ΑΦΚΟ και μετά θα προτείνω στη Γραμματεία να την κλείσει ως αναφορά. Το θέμα θα παραμείνει γιατί είναι ύψης της σημασίας. Τώρα φτάνουμε σε ένα άλλο θέμα. Αφορά τις απαιτήσει προσβασιμότητας. Η κυρία Κούνεβα είναι εδώ μαζί μας, που είναι η συγγήτρια. Κυρία Κούνεβα, έχετε το λόγο. Κάντε μας μια εισαγωγή επί του θέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι άνθρωποι με αναπηρία ενέρχονται σε 80 εκατομμύρια και καθώς η Ευρώπη γερνά, μέχρι το έτος 2020 οι άνθρωποι με προβλήματα αναπηρίας προβλέπεται να αυξηθούν σε 120 εκατομμύρια. Ακριβώς σε αυτό το λόγο Πιστεύω ότι το πρόβλημα της προσβασιμότητας δεν αφορά μόνο τους πολίτες με αναπηρίες, αλλά και τους ηλικιωμένους που αυξάνονται. Σε αυτό το σημείο του κειμένου που αφορά τον ορισμό του, ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι από την εφαρμογή της προτι... προτινόμενης οδηγίας, εισάγουμε την πρώτη μας τροπολογία. Πιστεύουμε ότι στους ωφελούμενους πρέπει να ενταχθούν όχι μόνο οι άνθρωποι με διαπιστωμένες αναπηρίες, αλλά και ηλικιωμένοι και όλοι όσοι εμποδίζονται στη κίνηση και επικοινωνία με το περιβάλλον. Επίσης, θα δείτε ότι προτείνουμε να μην χρησιμοποιείτε στο κείμενο η φράση πρόσωπα με λειτουργικού περιορισμού, καθώ είναι ένα όρο που ρίχνει ουσιαστικά στο άτομο την ευθύνη για την κατάσταση και τα εμπόδια του που συναντά. Επίσης, γνωρίζουμε και από τις αναφορές στην Επιτροπή ότι ενώ οι άνθρωποι με αναπηρίες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα κινητικότητας, προσβασιμότητας και απασχόληση, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν είτε δεν εφαρμόζονται, είτε το κάτι κράτος μέλος προσεκίζει την προβασιμότητα με διαφορετικές εθνικές οπτικές. Γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε και στον έλεγχο της νομοθεσίας που ήδη υπάρχει για την προβασιμότητα, αλλά και στην κάλυψη όλων των κενών εκεί που δεν υπάρχουν ούτε νόμοι ούτε αγωγή για την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους με αναπηρία, στους ηλικιωμένους και στα άλλα εμποδιζόμενα πρόσωπα. Ταξιδεύουμε συχνά και βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα σε κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να δεν τολμούν να περπατήσουν στους δρόμους για τον απλούστατο λόγο της απώλειας έλλειψης προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους, ηλικιωμένοι χαμηλού εισοδήματο, που μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ανάπερα παιδιά που δεν γίνονται αποτεχτά στα σχολεία. Γι' αυτό προτείνουμε και πιστεύουμε ότι η πρόταση για μια νέα οδηγία η οποία στοχεύει σε νέες διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσει προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα. Εάν αυτό το βήμα γίνει στη σωστή κατεύθυνση, με κριτήριο όχι μόνο της ανάγκης της αγοράς, αλλά και της ανάγκης της κοινωνίας, μπορεί να βελτιώσει τη ζωή όλων των εμποδιζόμενων ανθρώπων, να βοηθήσει τις οικογένειες των αναπήρων, στηρίζοντας την αρχή της ανεξάρτησης διαβίωση και να προσφέρει νέες δυνατότητες ανάπτυξης στην αγορά. Ο τίτλος της πρότασης του Συμβουλίου και της Κομισιόν κάνει λόγο για εννέες απαιτήσει προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Δηλαδή, για το πώς θα μπορέσουν όλοι οι πολίτες να χαρούν, να πλησιάζουν και να χρησιμοποιήσουν εύκολα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που βελτιώνουν τη ζωή μας. Και γιατί όχι, μας σώζουν από περιπέτειες επίσης. Παράδειγμα, ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο κινητό τηλέφωνο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος με προβλήματα όρασης σε μια περιοχή της Ελλάδας ή της Ιταλίας που κινδυνεύει από σεισμικές δονήσεις μπορεί να σώσει ακόμα και τη ζωή. Η πρόταση περιορίζεται αποκλειστικά μόνο σε καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες της ψηφιακής τεχνολογίας. Ειδικότερα η πρόταση αφορά ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λειτουργικά συστήματα, ATM και μηχανήματα έκδοσης εισιτήριων, smartphone, εξοπλισμό τηλεοράσεων, τηλεφωνικές υπηρεσίες, οπτικοακουστικές υπηρεσίες, ψηφιακές εγκαταστάσεις σε υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικό εμπόριο. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το πεδίο εφαρμογή αυτή τη πρόταση είναι πολύ περιορισμένο. Γι' αυτό και εμείς προτείνουμε δύο βασικές τροπολογίες. Πρώτη, να πλατείνουμε το πεδίο εφαρμογή της πρότασης με την προσθήκη νέων απαραίτητων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως μεταξύ άλλων είναι τα website, τα application, οι υπηρεσίες στέγασης σε νοσοκομεία και ξενοδοχεία, τα τερματικά πληρωμών, οι οικιακές συσκευές που λειτουργούν με διαπαφή χρήστη. Δεύτερη, να επιμείνουμε στη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά που λέμε δομημένο περιβάλλον. Δεν αρκεί να βρεις προϊόντα και υπηρεσίες προσβάσιμες. Πρέπει να μπορείς να φτάσεις κοντά τους. Αν δεν υπάρχει η μπάρα, το κατάλληλο σανσέρ για τον απρικό καρότσι ή η ειδική πρόσβαση για τον άνθρωπο με προβλήματα όρασης που θέλει να φτάσει στο ιατρείο ή το κατάλληλο προσωπικό πώς θα κατανοήσει τις δικές ανάγκες και τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου με νοητική στέρηση, τι νόηματα έχουν τα προσβάσιμα προϊόντα. Τι νόηματα έχει ένα προσβάσιμο ATM αν το εμποδιζόμενο πρόσωπο δεν μπορεί να προσεγγίσει το μηχάνημα και την είσοδο του τραπεζικού καταστήματος. Άρα, η προσβασιμότητα του δεμημένου περιβάλλοντος είναι το α και το ω. Τρίτη παρατήρηση. Επειδή το κόστος προσαρμογής των ψηφιακών προϊόντων είναι υψηλό, ιδιαίτερα σε μια ψηφική αγορά που κυριαρχείται στους τομείς της πατέντας από τις πολιτικές, πρέπει να εξετάσουμε τη μεγάλη προσοχή, τη μεγάλη προσοχή και να θέσουμε ασφαλιστικές δικλείδες ώστε το κόστος προσαρμογής να μην αυξήσει τη τιμή επιβαρύνοντας τις ευάλωτες κατηγορίες των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό το λόγο, αν θέλουμε να έχουμε μια αποτελεσματική οδηγία προσβασιμότητας, πρέπει να δώσουμε έμφαση στα εξή επίμαχα ζητήματα της πρότασης. Πρώτη, στις εθνικές αρχές υποπτίας, διότι αυτές πρέπει να ελέγχουν τη τήρηση της νομοθεσίας για την αναπηρία και την προσβασιμότητα εκεί που δεν υπάρχουν πρέπει να δημιουργηθούν. Δεύτερο, στη συμμετοχή των αντιπροσευτικών οργανώσεων αναπηρίας στη διαδικασία προετοιμασίας των εναρμονισμένων προτύπων, καθώς επίσης και στη συμμετοχή εκπροσώπων των εθνικών υποπτικών αρχών και των οργανώσεων στη, δημόσια, στη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας, η οποία θα μελετήσει τις καλές πρακτικές προσβασιμότητας. Τρίτο, επίσης δίνουμε μεγάλη σημασία στο ποιος, πότε και πώς θα κρίνει ή αν η προσαρμογή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας θα επιφέρει ανάλογη επιβάρηση αυτόν κατασκευαστεί εάν ζητήσει να εξαιρεθεί από αυτόν τον εννέο κανόνα προσβασιμότητας. Τέταρτο, στην ανάγκη να υπάρχουν κατανοητές εξηγήσει και αναλυτικές οδηγίες χρήσης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στην απαραίτητη κατάρτιση και επιμόρφωση των ανθρώπων. Πέμπτο, τελευταίο, στο χρόνο εφαρμογής της οδηγίας. Εκτιμάμε ότι τα έξι χρόνια μετά την έναρξη ισχύω της οδηγίας που θέτει ως χρονικό όριο η πρόταση για την εφαρμογή είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα για ψηφιακά προϊόντα που ανανεώνονται γρήγορα και έχουν όλα ένα και μικρότερο κύκλο ζωής προτείνουμε ο χρόνος για την εφαρμογή των μέτρων να μειωθεί ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας και του προϊόντος. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερα, σας ζητώ τη συμβολή σας έτσι ώστε από κοινού να συμβάλλουμε σε μια γνωμοδότηση άξιας και σημασίας που έχει αυτή τη σημαντική πρόταση οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνώ μαζί σας ότι το θέμα έχει ύψιστη ε, σημασία ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον πολιτισμό μας. Παρακαλώ συνάδελφοι, θέλετε να αντιδράσετε. Κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την πολύ καλή της δουλειά ήδη και για τις προτινόμενες τροπολογίες και το ε, σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, εμείς από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών καλωσορίζουμε τη σχετική ε, νομοθεσία, αυτή την πράξη για την προσβασιμότητα, διότι τα κράτη-μέλη έτσι θα κληθούν να σεβαστούν πλήρως τα δικαιώματα των ανθρώπων με κάποια αναπηρία και έτσι θα μπορέσει να υπάρξει κοινωνική και επαγγελματική ένταξη για αυτά τα άτομα και πλήρη συμμετοχή του στα κοινωνικά δρόμενα. Τώρα εμείς ως ε, ευρωβουλευτές θα πρέπει να φροντίσουμε το ε, πνεύμα και το γράμμα του νόμου να ταιριάζουν, να ταυτίζονται. Και αυτό έχει να κάνει και με το ρόλο της Επιτροπής Αναφορών άμεσα, που είναι πάντοτε να ε, βάζει σε πρώτο πλάνο τη φωνή του πολίτη και τις ανησυχίες του. Κατά την άποψή μας θα πρέπει πρώτα απ' όλα η δική μας Επιτροπή να εστιάσει στο σεβασμό του άρθρου 4.3 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Αυτή είναι η αρχή. Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς. Αυτό θα πει αυτό το άρθρο. Εμείς πρέπει να είμαστε οι φωνή, οι φωνές αυτών των ανθρώπων, των ανθρώπων με αναπηρία και θα πρέπει και οι οργανώσεις τους να ακουστούν και να βοηθήσουν στην ε, σύνταξη των ε, τροπολογιών. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δικές τους ανησυχίες, στις, στις τροπολογίες μας και ε, στις επαφές που θα έχουμε εντός και εκτός Κοινοβουλίου. Θέλω να σας πω ότι στην ακρόαση που είχαμε πέρσι τον Οκτώβριο, Είχαμε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις αναπηρίες ε, που εκπροσωπεί πολλά εκατομμύρια ανθρώπων με αναπηρία στην Ευρώπη. Τεράστιο, πολύτιμο το έργο αυτού του φόρουμ και πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δικές τους ανησυχίες και γνωρίζω έχοντας ακούσει τώρα την εισηγήτρια και τα σχολιά της και τις τροπολογίες ότι η εισηγήτρια ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και εμείς θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας. Δύο-τρία βασικά σημεία λοιπόν που θα ήθελα να επισημάνω. Ορισμένα συμφωνούν με τη θέση της εισηγήτριας, ε, κάποια ελαφρώς διαφέρουν. Πρώτα απ' όλα ο ορισμός ε, των ε, ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, τα εμποδιζόμενα πρόσωπα. Ε, σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, έχουμε μια γυράσκουσα κοινωνία, καλό είναι να έχουμε ένα πιο ευρύ ορισμό. Θα πρέπει βέβαια να εξασφαλίσουμε η νομοθεσία να συμπίπτει με την υφιστάμενη νομοθεσία, δηλαδή τους υφιστάμενους ορισμούς ε, σε ό,τι αφορά τι διάφορε μορφέ, μιλάμε για μειωμένη κινητικότητα, για παράδειγμα, limited mobility και έχουμε κάποιου ορισμού για τι αναπηρίε. Μην έχουμε διαφορετικού πολλάπλου ορισμού, γιατί έτσι μπορεί να δυσκολέψει τελικά η εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία. Τώρα, ε, γενικά συμφωνώ σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί τομεί που θα μπορούσε η πράξη αυτή να προχωρήσει περισσότερο, όπου υπάρχουν κενά, δημιουργούνται κενά και πιστεύω πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι όταν υπάρχουν κενά στην νομοθεσία, ε, όταν εμεί τα δημιουργούμε τώρα, θα τα λάβουμε στο τέλο από τη μορφή αναφορών. Θα μα γυρίσουν πίσω αυτά τα κενά. Επομένω, καλό είναι να μειώσουμε στο δυνατόν από τώρα αυτά τα κενά στην ε, νομοθεσία. Και καλό θα είναι ακριβώς όταν δούμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διάπονται από το νομοθεσία να φροντίσουμε να μην υπάρχουν και τέτοια κενά. Σε κάποιες περιπτώσεις και δίνω το παράδειγμα των μηχανημάτων ATM και των τραπεζών. Ε, εκεί έχουμε τους κανόνες νομοθεσίας που διέπουν αυτά τα μηχανήματα. Όμως ε, το σωματωμένο περιβάλλον ε, στη, στα ATM είναι ανοιχτό σε θελοντικά εθνικά μέτρα. Εκεί θα μπορούσε να δημιουργηθεί κενό. Δηλαδή, ναι, μεν είναι προσβάσιμο όταν φτάσεις εκεί, αλλά πώ θα φτάσει εκεί αν έχει ε, ένα ε, πρόβλημα, αν είσαι ένα εμποδιζόμενο πρόσωπο. Μπορεί να μην μπορεί να φτάσει εκεί. Και δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε αυτό το πρόβλημα που σα είπα, δηλαδή το πνεύμα και το γράμμα του νόμου τελικά να μην είναι ακριβώ το ίδιο. Τώρα, έρχομαι σε ένα άλλο θέμα, την έννοια του δυσανάλογου βάρου θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και συχνά μας υπενθυμίζεται με αλφαγιώτα ότι υπάρχει το πρόβλημα του διοικητικού βάρους, του κόστους, ε, της νομοθεσίας κτλ. κτλ και ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, για το κόστος, για τις βιομηχανίες κτλ. Όμως, εδώ βλέπω έναν κίνδυνο, πραγματικό κίνδυνο. Έχοντας έναν ορισμό δυσανάλογου βάρους, αλλά χωρίς να είναι σαφής ο ορισμός, τελικά δημιουργείται ένα παραθυράκι με την περίπτωση αυτή που θα μπορούσε κάποιο να το εκμεταλλευτεί και έτσι να μειωθούν τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων στην ομοθεσία. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες οι παράμετροι του ορισμού για το τι είναι υπερβολικά βαρύ. Ε, και τώρα, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, Πέντε χρόνια περιμέναμε να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτήν την πράξη. Την νομική είναι πολύ θετικό που τώρα την έχουμε εμεί. Αναχείρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάποιοι εδώ ζητούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρξει μια επικαιροποίηση ε, τη διαβούλευση του 2014 που θεωρείται κάπω παροχημένη, ξεπερασμένη. Εγώ θα έλεγα να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί έτσι θα μπορούσαμε να καθυστερήσουμε ακόμη περισσότερο τη διαδικασία και τελικά αυτά τα δικαιώματα ε, να αργήσουμε να τα εξασφαλίσουμε για αυτούς τους ανθρώπους που τόσο τα χρειάζονται. Είπε και η και συμφωνώ, πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε γρήγορα ε, την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, γιατί αν είναι πολύ μακρά αυτή η μεταβατική περίοδος, πολλά από τα προϊόντα και υπηρεσίες ε, θα έχουν εξελιχθεί πλέον και δεν θα καλύπτονται πια από το πεδίο εφαρμογή ομοθεσίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε μετά ε, και ποιο είναι το πραγματικό περιβάλλον. Και επανέρχομαι και στην προηγούμενη αναφορά με το διαδίκτυο, ότι η ψηφιακή κοινωνία και τα δικαιώματα που πρέπει να ακολουθούν τις ε, τεχνολογικές εξελίξεις στην κοινωνία. Άρα πρέπει και η περίοδος της μετάβασης να είναι η κατάλληλη. Τούτου λεχθέντος περιμένουμε φυσικά ε, να συνεργαστούμε πολύ καλά με την εισηγήτρια. Πρέπει η Επιτροπή Πέτη να τοποθετηθεί με μια σχηρή γνωμοδότηση για να ακουστούν οι φωνές αυτών που τόσο πολύ έχουν ε, μείνει μέχρι στιγμής ε, σιωπηλοί. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σντανόκα. Yes, θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο Κούνεβα για την εξαιρετική εργασία και για τη σωρία ε, προτάσεων καθώς και τροποποιήσεων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τον ορισμό. όπως φαίνεται στην τροπολογία 2 και σε άλλες τροπολογίες. Είναι μια πολύ καλή πρόταση και θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό το δεύτερο τμήμα, δηλαδή άτομα με αναπηρίες ή με ε, περιορισμούς και δυσλειτουργίες. Δεν θα πρέπει να γίνεται συσχετισμός, κάποιος ε, ηλικιακός συσχετισμός ή μία άλλη ε, διατύπωση γιατί μιλάμε για πληθώρα ανθρώπων που καλύπτει αυτός ο κανονισμός. Ε, δεν ξέρω ποια είναι ε, η άποψη ε, των άλλων εισηγητών, δηλαδή τι γνώμη έχει η αρμόδια επιτροπή. Μπορεί ενδεχομένως να μας το πει η κυρία Κούνεβα ποια είναι η άποψη της αρμόδιας επιτροπής. Νομίζω ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η εμβέλεια του κειμένου και ο κανονισμός θα πρέπει να ασχοληθεί και με άλλα συναφή ζητήματα. Δηλαδή δικαιώματα τα οποία ε, εντάσσονται σε προγενέστερες ε, σε προγενέστερα νομοθετήματα, νομοθετήματα, ιδιαίτερα σε σχέση με την τροπολογία 661 του 2009 και την συναφή τροπολογία. Γιατί ίσως υπάρχουν υπηρεσίες, αλλά η προσβασιμότητα είναι πολύ περιορισμένη. δηλαδή έμπρακτα υπάρχουν κενά στην ε, προσβασιμότητα. Και γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι λάβαμε μία σειρά αναφορών που δείχνουν ότι η προγενέστερη νομοθεσία δεν ήταν ικανή να λειτουργήσει όπως θα το επιθυμούσαμε. Επίσης, ως προς τροπολογία σας υπαριθμού 43, μιλάτε για την εισαγωγή ορισμένων ποσοστιαίων αναλογιών, δηλαδή προγραμμάτων, τα οποία θα πρέπει να έχουν ε, υποτιτλισμό και να προωθούνται και στην νοηματική γλώσσα Πώς ορίζεται αυτές τις ε, ποσοστιαίες αναλογίες. Ποια μπορεί να είναι η στάση μας ε, ως προς αυτή την πρόταση. Σε σχέση και με άλλους ε, φορείς που ασχολούνται με αυτό τον κανονισμό. Θα ήθελα να μου πει η εισηγήτρια Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής Απασχόλησης. Εγώ είμαι ε, σκιώδης εκεί και από όσο γνωρίζω έχουν περάσει δύο εβδομάδες πριν ορισμένα ε, θέματα. Επίσης, τροπολογία 65, αυτές οι χρονοθυρίδες εφαρμογής θα ήθελα να μου πείτε πώς τις αντιμετωπίζετε. Ελπίζω να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και κατά τη συνεργασία μεταξύ εισηγήτριας και σκιωδών για το τελευταίο τελικό κείμενο γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή είχαμε πολλές ερωτήσεις, θα δώσω το λόγο και πάλι στην κυρία Κούνεβα στο τέλος, αλλά θα ήθελα η Επιτροπή να λάβει το λόγο πριν. Σας ευχαριστώ. Okay, that's, that's okay. <laughs> Έκανα λάθος και σας προσφώνησα ως κύριο, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. Ε, κυρία μου λοιπόν, ε, παρακαλώ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη γιατί αργήσαμε, δεν φταίγαμε, αλλά δεν καταλάβαμε καλά τα ωράρια. Επήξε κάποια παρανόηση και λυπούμαστε πολύ αλλά δεν ήμασταν από την αρχή, χάσαμε λίγα λεπτά. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για το σχέδιο γνωμοδότησης. Είναι πολύ αναλυτικό, άρτιο, λεπτομεριακό και με πολύ χαρά σημειώνουμε ότι στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό είναι σημαντικό γιατί το έγγραφο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία αλλά και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία εν γέννη. Σημειώνουμε επίσης την επιθυμία της εισηγήτριας ε, να υπάρξουν περισσότεροι τομεί παρέμβαση, δηλαδή να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας ε, και σίγουρα οι προτάσεις ε, θα αποτελέσουν αντικείμενο μια σοβαρής σημαντικής συζήτησης εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις. Διαβάζοντας το σχέδιο γνωμοδότησης, πρέπει να πω ότι ε, μας δημιουργήθηκαν κάποιες απορίες, ε, κάποιες θετικές, κάποιες λιγότερο, παραδείγματος χάρη σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για αυτές τις λειτουργικές απαιτήσει. Δηλαδή να έχουμε παραπάνω ορισμούς, ε, περισσότερες επεξηγήσεις. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για την καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής της οδηγίας, οπότε φαντάζομαι ότι ε, θα μπορούσαν σε αυτές τις προτάσεις να περιληφθούν πολύ χρήσιμα πράγματα για να είναι πιο ευνόητη και ευεφάρμοστη η πρόταση οδηγίας. Λίγο λιγότερο ε, συμφωνούμε με το να βάλουμε του εμποδιζόμενου και τους ανθρώπους με αναπηρία στο ίδιο επίπεδο ακριβώ. Στην πρόταση οδηγία. λέμε ότι ό,τι θα γίνει για τα άτομα με αναπηρία θα μπορούσε να είναι χρήσιμο να αποδώσει καρπούς και για άτομα με κάποιους περιορισμού, ε, ε, για εμποδιζόμενα πρόσωπα, αλλά είναι πολύ ευρύ ορισμό του εμποδιζόμενου προσώπου και κάπως ε, ίσως αυθαίρετος κάποιες φορές. Ε, δεν θέλουμε να ανοίξει πάρα πολύ το πεδίο εφαρμογής ε, της οδηγίας και να καλύψει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού που δεν είναι μόνο το πρόβλημα η ποσότητα, αλλά το, θα είναι δύσκολο να ορίσουμε τι ακριβώς, ποιες ακριβώς κατηγορίες προσώπου περιλαμβάνονται Νομίζουμε ότι η προσέγγιση μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πιο ε, ισορροπημένη. Είπαμε δηλαδή ότι ό,τι κάνουμε για τα άτομα με αναπηρία θα μπορεί να χρησιμεύσει, θα είναι χρήσιμα και για τα άτομα τα εμποδιζόμενα. Αλλά να μην αφομοιώσουμε το ένα με το άλλο ε, γιατί νομίζουμε ότι αυτό στην πράξη θα μπορούμε να το διαχειριστούμε πολύ δύσκολα. Επίσης έχουμε κάποιες απορίες και κάποιες ερωτήσεις σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη τη διαφορετική προσέγγιση για την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας ανάλογα με την υπηρεσία, ανάλογα με το προϊόν. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η προθεσμία των 6 ετών ε, θεωρείται ότι είναι μεγάλη και ότι δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να υπάρχει εξαετία για όλα τα προϊόντα. Εμείς όμως θέλουμε να είναι απλό, να είναι βανάγνωστο, να είναι εύληπτο για τον καταναλωτή, για τις επιχειρήσεις και για τις διοικήσεις ε, των κρατών μελών. Μια διαφορετική λοιπόν από ε, προσέγγιση. Ανάλογα με την ή ανάλογα με το προϊόν, θα μπορούσε κατά την άποψή μα να οδηγήσει σε σύγχυση. Επίση, ε, δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ω προ το, τη δική μας πρόταση για την ε, εξαιρέσεις κοινοποίηση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που μας είναι πολύ απαραίτητες ε, από οικονομικής πλευράς. Εδώ μιλάμε μόνο για την κοινοποίηση βέβαια. Αυτό το σημείο βλέπουμε να ε, λείπει από την πρόταση. Θα υπήρχε σίγουρα ένας μεγάλος οικονομικός αντίκτυπος και μεγάλο διοικητικό βάρος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι μονοπρόσωπες ή να έχουν δύο άτομα. Σίγουρα θα είναι μεγάλο το διοικητικό βάρος. Ε, πάντως σημειώνουμε πολύ ενδιαφέρον τις ε, προτάσεις αυτές για συμπληρωματικούς ορισμούς ε, που θα κάνουν πιο ξεκάθαρο το κείμενο. Και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ληφθεί καλύτερα υπόψη το feedback τι έχουν να μας πούν οι ενώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία που πραγματικά έχουν εμπειρία και είναι πάρα πολύ χρήσιμη και η τεχνογνωσία τους και η εμπειρία τους και μπορούν να βοηθήσουν και τις ε, εποπτικές αρχές και την Κομισιόν. Αυτό το διάλογο άλλωστε τον έχουμε ήδη ξεκινήσει και θα συνεχίσουμε ε, στον ίδιο δρόμο. Πολύ επικοδομητική πάντως αυτή η ιδέα ε, νομίζουμε ότι θα επιτρέψει ε, μία όσο το δυνατόν ε, πιο ρεαλιστική ε, αποδοτική εφαρμογή της οδηγίας. Δεν ήθελα να δαπανίσω πολύ από το χρόνο σας. Έκανα κάποιες γενικές παρατηρήσεις μόνο πάνω σε ένα πάρα πολύ αναλυτικό, πληρέστατο κείμενο. Σας έδωσα κάποια στοιχεία. Πρέπει να πω ότι χαιρόμαστε πολύ που έχουμε μία τόσο θετική ανταπόκριση στις δικές μας προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους. Να σας πω ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί φυσικά. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 29 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και θα ψηφίσουμε κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης εδώ στην Επιτροπή μας τον Ιανουάριο. Να ευχαριστήσω την κυρία Κούνεβα και βεβαίως έχετε το λόγο. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις παρατηρήσεις σας. Ε, θα σας πω σύντομα κάποιες σκέψεις. Ο ορισμός πρέπει να μην εξαιρεί κανένα από τα εμποδιζόμενα άτομα. Θα δουλέψουμε μαζί για να καταλήξουμε στον καταλληλότερο ορισμό ε, έχω, έχω και εγώ μια απορία ακριβώς τι θα επιλέξουμε. Γιατί και εγώ ήδη είμαι ένας άνθρωπος με διάφορα προβλήματα και με πολύ βαρύ αναπηρία. Και νομίζω ότι είμαι πολύ χρήσιμη σε αυτό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε και το ορισμό και ολόκληρη την έκθεση. Συμφωνώ με την κυρία Ντάρλινγκ για, ε, για τους φόβους της, ε, σχετικά με το δυσανάλογο βάρος και τόσο και με πολλές από τις παρατηρήσεις σας και πιστεύω ότι τα κάνουμε πολύ καλή δουλειά ως Επιτροπή και ότι τα συνεργαστούμε άριστα. Επίσης, να, να πω στην κυρία Σντάνουκα ότι η αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικής Αγοράς δεν έχει ορίσει ακόμα το τελικό εισηγητή ή πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή στο πρόσωπο και έτσι δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωμένη άποψη για την γνώμη της Επιτροπής. Ε, για τις απόψεις δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω γιατί είχαμε μόνο μια ακρόαση επί του θέματος στην Επιτροπή. Τα τεχνικά ζητήματα, τα ποσοστά, επιφυλάσσομαι να σας απαντήσω αναλυτικότερα. Θέλω να σας πω ότι τα τεχνικά ζητήματα, τους ορισμούς, συζητήσαμε πολύ με τους οργανώσεις και τους εμπειρογνώμοντες. Αλλά όπως φαίνεται υπάρχουν αρεύματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε και να βρούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ε, Το ίδιο ισχύει και τις ημερομηνίες. Επίσης με προσοχή βλέπουμε τα ζητήματα των μικρών επιχειρήσεων και την εξαίρεση κοινοποίηση επιφυλάσσουμε. το κατατέσσουμε και τροπολογίες και νομίζω η συνεργασία μας, η συνεργασία μας θα εξελίξει την έκθεση αυτή σε ένα καλό κείμενο. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να επαναλάβω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 27η Οκτωβρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και τώρα πάμε στην επόμενη έκθεση στην ημερήσια διάταξή μας για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών το 2015 ο συνάδελφο Βαλίνα είναι. Ε, Βαλίνα είναι η συγγήτρια. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το σχέδιο της ετήσιας έκθεσης τη επιτροπή Αναφορών για το 2015, για το οποίο λάβαμε 1.431 αναφορές. Αυτό συνιστά μείωση κατά 46% σε σχέση με το 2014. Από αυτές 424 αναφορές εξετάστηκαν ε, και αιτήσαν. 519 είναι ανοιχτές και 483 κρίθηκαν μη παραδεκτές. Μέσω αυτής της ετήσιας έκθεσης ε, η Επιτροπή μας ε, ουσιαστικά παρακολουθεί τα σημαντικότερα γεγονότα της προηγούμενης χρονιάς και επίσης αναφέρει την άποψή της για τη λειτουργία της Επιτροπής, τη σχέση της ε, με τα άλλα θεσμικά όργανα και φυσικά κυρίως με τους πολίτες μας που πρέπει να είναι στο επίκεντρο όχι μόνο της δικής μας Επιτροπής αλλά και όλων των ευρωπαϊκών διοικήσεων. Θα είμαι σύντομη, δεν θα επεκταθώ πολύ σε λεπτομέρειες διότι ήδη έχετε όλοι και όλες την έκθεση αυτή. Θα ήθελα πάντως ε, να τονίσω το ότι όπως είδαμε και το βλέπουμε ακόμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις Έχουμε την ανθρωπιστική κρίση των προσφύγων. Έχουμε θανάτους ε, εκατοντάδων μεταναστών στις πόρτες ε, της Ευρώπης. Έχουμε τη βία, τις ανισότητες ε, μεταξύ των φίλων, την αύξηση της ξενοφοβίας, ε, την πολύ ε, μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση που πλήττει τους πιο φτωχούς και συνεχίζουν να χάνονται τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Σας είπα λοιπόν ότι είχαμε 1431 αναφορές το 2015 και κυρίως έχουν ως αντικείμενο αυτά τα θέματα, αλλά και άλλα όπως είναι οι αναπηρίες ή το περιβάλλον. Επίσης σχεδόν πάντοτε αυτές οι αναφορές απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τελικά είναι και ο θεματοφύλακας ε, τον, ε, για την τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων και γι' αυτό στο πλαίσιο της έκθεσης θέλω να εκφράσω το ότι πολλές φορές η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δείχνει το απαραίτητο ενδιαφέρον για να απαντά ε, με το δέοντα τρόπο στις αναφορές. Νομίζω ότι το δικαίωμα υποβολής αναφορών θα πρέπει να είναι ένας από τους μηχανισμούς για τη βελτίωση της ζωής των προσώπων, να περιορίζει τις αποστάσεις μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών διοικήσεων. Γι' αυτό είναι σημαντικό ε, να διατεθούν περισσότεροι πόροι και τεχνικοί και ανθρώπινοι στην Επιτροπή μας. Επίσης είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει το ρόλο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών των πολιτών με βάση τις, ε, τις συστάσεις που έκαναν οι οργανώτες των πρωτοβουλίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ξέρουμε, παραδείγματο χάρη, τι έγινε με την πρωτοβουλία για το δικαίωμα στο νερό. Απολύτω τίποτα. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δική μα η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται. Εμεί θέλουμε να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τι αναφορέ ε, για να δώσουμε στη δημοσιότητα τι τραγωδίε, τι σημαντικότερε τραγωδίε και δράματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ. Παραδείγματο χάρη, στην Ολομέλη συζητήσαμε την νομοθεσία για τα στεγαστικά δάνεια, χρηματοοικονομικά άλλα εργαλεία, προτιμησιακά δάνεια, αυτά δηλαδή που πρέπει να εξοφληθούν κατά προτάτη και τα λοιπά. Ξέρουμε ότι τουλάχιστον στη χώρα μου, την Ισπανία, έμειναν εκατοντάδε οικογένειε σε κατάσταση μεγάλη φτώχεια ε, λόγω υπερχρέωση. Επίση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ε, ότι έχουμε και ένα ρόλο σύνδεση με το διαμεσολαβητή. Ε, στην περίπτωση τη διαμεσολαβήτρια και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Πολίτη, με ε, την ε, διαμεσολαβήτρια που είπε ότι θα πρέπει να δουλέψει σοβαρά, καταδικάζει τις περιστρεφόμενες πόρτες, έχουμε το έργο της Frontex. Τέλος πάντων θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε εδώ όχι απλά την εκπαιρέωση και κλείσιμο αναφορών, αλλά να βοηθήσουμε πραγματικά τους πολίτες της Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, θέλει κάποιος το λόγο. Αν όχι, Εγώ ως σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ ε, και όχι ως πρόεδρος να σας ε, συγχαρώ για την έκθεση. Πραγματικά αποτελεί μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Εκτιμώ τις θέσεις σας σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ε, ιστοσελίδας. Είναι πολύ καλή η ιδέα σας να εμπλέξουμε περισσότερο τα κράτη-μέλη σε αυτή τη διαδικασία και βεβαίως να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και με άλλες επιτροπές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά. Οπότε θα ε, υποβληθούν κάποιες τροπολογίες, αλλά ε, η βάση πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Η κυρία Σιμάνσκι τώρα έχει το λόγο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Αξιότιμα μέλη. Διάβασα την έκθεση, το σχέδιο έκθεση της κυρίας Βαλίνα με πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως ε, ε, υπεύθυνη για την ε, διάδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Επιτροπή σας. Συμφωνώ με τις απόψεις που εκφέρονται στην έκθεση ότι υπάρχει στενή εργασιακή σχέση μεταξύ της Επιτροπής σας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή ακριβώς η στενή συνεργασία είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε ότι οι αναφορές θα την χάνουν της προσοχής που τους αρμόζει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι ουδέτερος εταίρος, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τις σοβαρότητα των αναφορών και εμπλέκεται στην όλη διαδικασία. Επιβεβαιώθηκε από τον πρώτο αντιπρόεδρο, κύριο Τίμερμαν, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του τον Απρίλιο εδώ στην Επιτροπή σα. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει λεπτομερείς απαντήσεις στις, ε, στα αιτήματα για ενημέρωση από την Επιτροπή σας, όπου η αναφορά εμπίπτει στις αρμοδιότητες βεβαίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης πάντα έχει στόχο να εξασφαλίζει ότι στέλνει τους πιο αρμόδιους υπαλλήλου τη για να ε, παρέμβω στη συζήτηση για τα θέματα που ε, ασχολείται η Επιτροπή σα. Επίση, προσπαθούμε να παράσχουμε στην Επιτροπή σα ε, ουσιώδε απαντήσει και να το κάνουμε αυτό έγκαιρα. Που σημαίνει εντό των προθεσμιών που μα τίθενται. Ε, για το σκοπό αυτό και σύμφωνα και με τι δεσμεύσει που ανέλαβε ο ε, πρώτος αντιπρόεδρος Τίμερμαν στις 19 Απριλίου του τρέχοντος έστειλε μια επιστολή στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που ζητά από τα κράτη-μέλη να μειώσουν τις, ε, τους χρόνους απάντησης στα ίδια αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βοήθεια και για πληροφορίες για θέματα που άπτονται των αναφορών. Όπως ξέρουμε όλοι, πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ζητήσει από τα κράτη-μέλη ενημέρωση. Οπότε, κλείνοντας να πω ότι ο πρώτος αντιπρόεδρος, Τίμερμανς, βεβαίως θα αναφερθεί σε όλα τα θέματα, σε όλα τα ερωτήματα που σας απασχολούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια και βεβαίως προσβλέπουμε στην συνέχεια της πολύ καλής συνεργασίας που είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Να υπογραμμίσω απλώ στου ε, συναδέλφου ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 21η Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή της 29ης Νοεμβρίου. Η κυρία Βαλίνα για να ακούσουμε τα τελικά της σχόλια. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και για τα δικά σας σχόλια, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας και αν θέλετε μπορούμε να συναντηθούμε για τροπολογίες συμβιβασμού και να συνεργαστούμε έτσι ώστε αυτή η έκθεση να αφορά όλους και όλους. Κυρίες και κύριοι, Φαίνεται ότι τελειώνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Σας εύχομαι καλό βράδυ και θα συνεχίσουμε εδώ αύριο στις 9 το πρωί. Γεια σας.